Ε, με τις δηλώσεις τους για την διεθνή προστασία των καταγγελόντων. Don't worry, I know very well your job. <laughs> Sorry. I welcome this. Χαίρομαι που έχω ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε την ε, διεθνή προστασία των ε, καταγγελόντων μετά τη συζήτηση που είχε η Επιτροπής Γιώροβα μαζί σας πριν από 10 μήνες. Βεβαίω απαιτείται ένα ιδιαίτερο θάρρος για να καταγγείλει κανείς ε, κάποιες πρακτικές όπως η διαφθορά και βεβαίως είναι και θέμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ε, ελευθερίας της πληροφόρησης. Και όπως αναφέρθηκε και στην συζήτηση για το θέμα αυτό τον Απρίλιο που μας πέρασε, δεν υπάρχει ένα εναρμονισμένο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των κατακελώντων και η Κομισιόν γνωρίζει πως το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πολλές φορές να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα όπως πολύ καλά γνωρίζετε στην περίπτωση στην οποία δεν υπάρχει κάποιο ειδικό κλαδικό ευρωπαϊκό δίκαιο επαφίεται στα κράτη-μέλη να ρυθμίσουν το ζήτημα. Η Κομισιόν παρακολουθεί την νομολογία του ε, ΕΔΑΔ ε, και τις ε, συζητήσεις που γίνονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μια πιθανή συνθήκη πλαίσιο. Είχαμε και τις συστάσεις του 2014 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία καταγγελόντων που ζητούν από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να δημιουργήσουν ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία τους και η Κομισιόν καλωσορίζει το ότι πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο σε κάποια κράτη-μέλη. Να σας πενθυμίσω επίσης πως η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεβλήματος χρήματος του 2014 περιέχει κάποιες διατάξεις για την προστασία όσων αναφέρουν ύποπτες ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Επίσης τον ε, Δεκέμβριο πέρσι η Κομισιόν υιοθέτησε μια εφαρμοστική οδηγία για τον κανονισμό κατάχρησης ε, δεσπόζουσας θέσης για να προστατεύσουμε τα άτομα εκείνα τα οποία αναφέρουν παραβιάσεις του κανονισμού. Επίση, θα θυμάστε πω το Δεκέμβριο πέρσι εσείς εγκρίνατε μια οδηγία για την προστασία εμπορικών μυστικών ε, από την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψή τους και εκεί πέρα ενισχύθηκαν τα δικαιώματα των καταγγελόντων. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία οποιοδήποτε μιλάει για παρανομή απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη τέτοιων μυστικών θα απορρίπτεται εάν αποκαλύπτεται με την αποκάλυψη αυτή κάποια παρανομία ή δραστηριότητα που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον. Υπάρχει επίσης και η εκθέση του 2013 για την διαφθορά που αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Σημαντικά λοιπόν ζητήματα στις ε, συζητήσεις μας με τα κράτη-μέλη. Τέλος, η Κομισιόν θέλει να διασφαλίσει ότι οι καταγγέλλοντες που καταγγέλουν τέτοιες περιπτώσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα δημιουργηθεί θα χάνουν τις προστασίας που προβλέπει το Εθνικό Δίκαιο. Όπως ξέρετε, η υπόθεση αυτή συνεχίζεται και θα εκτιμούσαμε βεβαίω και την στήριξη του Κοινοβουλίου στη σύσταση αυτή τη υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, για να συνοψίσω, πολλά έχουν ήδη γίνει στο ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί όπου έχουμε αρμοδιότητα. Η Κομισιόν παρακολουθεί τι εξελίξει για να αξιολογήσει την πιθανή ανάγκη περαιτέρω δράση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα με χαρά θα ακούσω τις δικές σας απόψεις για το πώς μπορεί αυτή η δράση να βελτιώσει την προστασία των καταγγελώνων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Commissioner. το Ευρωπαϊκό σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την δήλωση που έκανε για το θέμα αυτό. Επί της αρχής είναι θετικό το ότι συζητάμε αυτό το θέμα για το πώς δηλαδή θα καταλήξουμε σε μια λογική αντιμετώπιση του θέματος και ειδικά στο θέμα του πού ακριβώς βρίσκονται τα όρια, γιατί καμιά φορά θεωρούμε τους καταγγέλλοντες ε, ως φάρμακο διαπασανώσεων. Να πω εδώ πέρα πως ε, εμείς ε, στο ΕΛΚ δεν είμαστε υπέρ μιας γενικής προστασίας η οποία θα κατσχύει και του ποινικού δικαίου. Μια λογική διαδικασία βεβαίως θα μας έβρισκε σύμφωνους. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις δομές, δομές εντός των επιχειρήσεων και των αρχών, έτσι ώστε σε πιθανές ε, παρανομίες οι οποίες αποκαλύπτονται να υπάρχει η ανάλογη προστασία. Η συζήτηση βεβαίως είναι περίπλοκη και δύσκολη γιατί περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς ελευθερία της γνώμης, ε, ιδιωτική ζωή, εθνική ασφάλεια, επιχειρηματικά μυστικά, απάτη και πιθανώς και φορολογικά ζητήματα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να κρίνουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Δεν μπορεί να τα βάζουμε όλα μαζί σε ένα κουβά και να λέμε προστατεύουμε γενικώ και αδιακρίτως. Θα πρέπει να διακρίνουμε τους διάφορους τομείς και περιπτώσεις και θεωρούμε πως ε, τελικά αυτή η προστασία είναι μια εθνική υπόθεση και αρμοδιότητα. και μπορούμε βεβαίως να ανταλλάξουμε κάποιες κατευθύνες γραμμές ε, και οδηγίες αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή του κράτους δικαίου η οποία θα πρέπει να είναι σεβαστή. Σας ευχαριστώ. Κύριος Λόπες Αγγιλάρ από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε. Γιατί μιλάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε για ένα πολύ επικαιρό θέμα και πολύ σοβαρό θέμα. Ε, γύρει πολλές ανησυχίες. Η προστασία των θεμελιών δων ε, δικαιωμάτων των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Και η προστασία αυτό, αυτών που λέμε στα αγγλικά whistleblowers, των καταγγελόντων. μιλάμε για άτομα τα οποία καταγγέλουν, ας πούμε, περιπτώσεις διαφθοράς, απάτες, οικονομικά, ε, οικονομική διαφθορά. Ε, επομένως, δηλαδή, ε, συνεργάζονται με διάφορες διοκτικές αρχές αυτοί οι άνθρωποι για να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά. Ξέρετε την περίπτωση Snowden, όπου υπήρξαν κάποιες πολύ δυσδυτικές πρακτικές που διέβρωναν τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά όλων των πολιτών από την ε, National Security Agency, την Αμερικάνικη. Μιλάμε λοιπόν για την ανάγκη να προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που καταγγέλουν, ε, που, που ενημερώνουν την ε, δικαιοσύνη για οικονομικές απάτες, για οικονομικούς και φορολογικούς παραδείσους, για εγκλήματα κάτω του περιβάλλοντος, της υγείας κτλ. Νομίζω ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να εγγύθουμε τα ε, δικαιώματά Το 2013 εγώ είμαι σε μια επιτροπή που ασχολούμαστε με τα, τις μαζικές ε, παρακολουθήσεις ε, στην Επιτροπή δηλαδή ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Κάναμε μάλιστα και τότε μία ακρόαση στην Επιτροπή αυτή δικαιοσύνη για να υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας ούτω ώστε με βάση το άρθρο 11 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα. Ε, ώστε αυτά που κάνουμε εμείς να συνάδουν και με αυτά που λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και κυρίως για να εξασφαλίσουμε τη μυστικότητα ε, αυτών των ανθρώπων που καταγγέλουν. Ε, να, πώς θα προστατεύσουμε καλύτερα τα άτομα αυτά με μια ομοιόμορφη ευρωπαϊκή νομοθεσία σύμφωνα με τις ε, εντολές ε, στις οποίες ε, και στα πορίσματα στα οποία κατέληξε η ε, Επιτροπή στην οποία εγώ προείδρευα. Αυτά έπρεπε να κάνουμε και πρέπει να τα υλοποιήσουμε τώρα. Τόμασιτς, από τους Ευρωπαίους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ. Ο ρόλος των καταγγελόντων είναι πολύ σημαντικός για κάθε κοινωνία είναι άτομα με ιδιαίτερο θάρρος και υπευθυνότητα που μας προειδοποιούν για ένα ζήτημα πριν αυτό γίνει άλυτο. Πρέπει λοιπόν να τους αναγνωρίζουμε για τη βοήθειά τους αυτή, παρόλο που πολλές φορές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους μετά από λίγο καιρό. Υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα και διαφθορά και οι κατακέλλοντες δυστυχώς δεν αποζημιώνονται ποτέ. Σε πολλές αναπτυγμένες χώρες δεν μπορούν καν να ε, βρούνε τους καλούς δικηγόρους γιατί οι δικηγόροι αυτοί είναι υπάλληλοι μεγάλων ε, εταιριών που είναι πλεγμένες αυτά. Οπότε βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν πιο επικοδομητικά τους καταγγέλλοντες, διότι ακριβώς οι καταγγέλλοντες είναι αυτοί που μας καταδεικνύουν τι πρέπει να αλλάξουμε σε μια κατάσταση και επειδή ξέρουν τα πράγματα από μέσα μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά. Γι' αυτό να προωθήσουμε το θετικό ρόλο των ατόμων αυτών στις κοινωνίες μας και χώρες μας πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να υπάρξει νομική αρρωγή να πάσα στιγμή προς αυτούς. Αλλά και οι καταγγέλλοντες από τρίτες χώρες επίσης πρέπει να προστατεύονται με άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύονται και αυτοί και οι οικογένειές τους από πράξεις εκδίκησης και ίσως και από δολοφονία. η κυρία Ρουίθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τον κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ, ναι, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο προστασίας. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να ανακαλύψουμε εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία αλλιώ πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσαμε να είχαμε αποκαλύψει. Όταν εγκλήματα γίνονται από μεγάλες εταιρείες, συνεταιρισμούς κτλ είτε από πολιτικού στα πλαίσια των κομμάτων του σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο να του επιβληθούν κυρώσει. Οπότε οι είναι το στοιχείο κλειδί για να αποφύγουμε την ατιμορρησία. Η σύμβαση κατά τη διαφθορά που ισχύει από το 2005 και που έχουν επικυρώσει ήδη μερικέ χώρε, αναγνωρίζει το ζήτημα. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να μην έχουν προστασία καταγγέλλοντες σε πολλές περιπτώσεις παραμένουμε σε δηλώσεις. Ναι, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ευαίσθητο το ζήτημα. Μόνο τέσσερι χώρε μέλη έχουν πάντω εκτενή νομοθεσία για την προστασία των καταλακιόντων. Πρέπει να υπάρχει μια νοοτροπία προστασία και να υπάρξει κατάλληλη νομοθεσία προστασία των ατόμων αυτών. Στην Ισπανία βρισκόμαστε πολύ πίσω, όπω και πολλέ άλλε χώρε βέβαια. Και σα διαβεβαιώ ότι θα είχαμε πολύ λιγότερη διαφθορά αν είχαμε καλή νομοθεσία για την προστασία των καταγγελόντων. Σίγουρα χρειάζεται ένα νομικό καθεστώς. Όταν κάποιος παίρνει την απόφαση να τολμήσει, να καταγγείλει ένα σοβαρό αδίκημα, είτε σε κόμμα είτε σε τέτοιο οτιδήποτε, πρέπει να προστατεύεται η ανωνυμία του και δεν πρέπει να κινδυνεύει ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του. Χρειάζονται τα άτομα αυτά προστασία για τη φυσική τους ακαιρεότητα πρώτα απ' όλα. Να υπάρχουν λοιπόν συμφωνίες για τέτοιες περιπτώσεις καταγγελιών. Να υπάρχει νομική αρρωγή δωρεάν για αυτούς. Να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ψυχολογική βοήθεια εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Γιατί εδώ μιλάμε για άτομα τα οποία δέχονται φοβέρες επιθέσεις που θέλουν να τους εκμηδενήσουν εντελώς. Και όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν και σε διεθνές επίπεδο και το Julian Assange τα γνωρίζουμε. Η ομάδα εργασία λοιπόν τη ΥΠΑ τη Αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΕΕ κατέληξε στο ότι αυθαίρετα ε, βρίσκεται σε Όλοι λοιπόν, Πρόεδρε, πρέπει να φροντίσουμε να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και χρειάζεται ένα νομικό πλαίσιο προστασίας των ατόμων αυτών. Ευχαριστούμε. Υπάρχει για σας μπλε κάρτα. Θέλετε να ακούσετε και να απαντήσετε. Παρακαλώ, κύριος Τζέιμς έχει την ερώτηση. Ή κύριε συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ που δέχεστε την ερώτησή μου. πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας. Αναφερθήκατε σε επιχειρήσεις, σε εταιρείε. Θέλω να το διασταυρώσω αυτό με σας. Εσείς λέτε ότι μόνο εταιρείε, επιχειρήσεις θα είναι το αντικείμενο της ρύθμισης αυτής την οποία ονειρεύεστε και πολιτικές οργανώσεις, χώρες, τοπικές αρχές, οποιαδήποτε οργάνωση θα μπορούσε να, να καταγγελθεί από ένα τέτοιο άτομο. Οπότε εγώ δεν βλέπω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό να το επηρεάσει. Αλλά περιμένω να μου απαντήσετε. Απάντηση. Ναι. Λοιπόν, Πρόκειται για δικήματα πολύ ειδικά συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά, έχουν να κάνουν με εγκλήματα ιδιαίτερα περίπλοκα, τα οποία λαμβάνουν χώρα μέσα σε χώρους που είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Συνεπώς η νομοθεσία, μέρος της τουλάχιστον, πρέπει να είναι εθνικό, αλλά πρέπει να υπάρχουν και διατάξεις κοινοτικού χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα γιατί δεν έχουμε δουλέψει αρκετά πέρα από τις συμβάσει, πέρα από τα θέματα που έχουμε αναπτύξει εδώ, τα είπε και ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ και οι χώρες μέλη δεν έχουν προχωρήσει. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί μέρος των αδικημάτων αυτών που παραμένουν ατιμόρυτα είναι σε αυτό το πλαίσιο αδικήματα πολυεθνικών ή κρατών ή πολιτικών κομμάτων. Τα γνωρίζουμε και στη δικιά μου τη χώρα τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτά και ευχαρίστως να μιλήσω μαζί σας για να δούμε τι πρέπει να γίνει μαζί. Από την ΚΟΕ, το λόγο έχει Κρέσπο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, η Wikileaks, Λίστα Λουξ Λίξ, Chelsea χάρη στη δράση των καταγγελόντων ή των υπερασπιστών του δικαιώματος στην ε, πληροφόρηση, η διεθνής του ε, δικαιωματο γνώμη γνώρισε ότι, μεταξύ άλλων, ότι οι Αμερικανικές αρχές ε, πίεσαν τις Ισπανικές κυβερνήσεις και άλλες για να κρύψουν στοιχεία για τα βασανιστήρια της CIA. Ο Χωσέ Κάουσο, δημοσιογράφος ε, προσπάθησε να μιλήσει για το τι έκαναν οι Αμερικανικοί, ε, ο Αμερικανικός στρατός στο Ιράκ. Μιλάμε για ε, κατασκοπή ευρεία κλίμακα, μιλάμε για περιπτώσει απάτη κτλ. Μιλάμε για φοβερά εγκλήματα. Και οι άνθρωποι που τα καταγγέλνουν θα πρέπει να θεωρηθούν υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ω μια ομάδα ιδιαίτερα ευάλωτη που απαιτεί ιδιαίτερη ε, προστασία. Και χαίρομαι που διάφοροι που μίλησαν εδώ σε, αυτό, σε αυτή την αίθουσα προς αυτή την κατεύθυνση ε, κινήθηκαν και μιλήσαν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπιστεί αυτά τα άτομα, ε, τα οποία υπερασπίζονται και καταγγέλ, καταγγέλλοντας περιπτώσεις διαφθοράς. Αν δεν έχει κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δύο λοιπόν ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες έχω να πω. Τι, θα, τι προβλέπετε νομοθετικά ε, εσείς ε, κομισιόν τους επόμενους μήνες για να προστατεύσετε αυτά τα άτομα. Θα θέλαμε επίσης να μάθουμε τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, άποψη του ΟΗΕ για τις παράνομες κρατήσεις του Χούλιαν Ασάνς που επί χρόνια κρατείται στην πρεσβεία του Εκουαδό στο Λονδίνο τι θα μπορέσετε να κάνετε ούτως ώστε να επιληθεί το θέμα του Ασάνς. Είναι πολύ συγκεκριμένες αυτές οι ερωτήσεις. Από τους πράσινους, ο κύριος Γιάβορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Άντερ Τούρκη, Στρακ, Άντρας Χόρβατ και πολλά άλλα ονόματα θα μπορούσα να σας πω. Δεν είναι ονόματα απλά κάποιων ανθρώπων, είναι μοίρες ανθρώπων οι οποίοι ανέφεραν πράγματα, περιστάσεις όπου κινδύνευε το δημόσιο συμφέρον και δεν υπήρξε καμία διαδικασία μάλλον υπήρχαν μόνο δίκες εις ε, βάρος τους. Εταιρείε και οι αρχές ε, τους επιτέθηκαν. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη να υπάρχει ένα καθεστώς προστασίας για, τον ανθρώπο, για τους ανθρώπους οι οποίοι ε, αποκαλύπτουν πληροφορίες. Πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή οδηγία και τα κράτη-μέλη να έχουν κάποια ελάχιστα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σέβονται όλα. Και βεβαίως η προστασία αυτή θα πρέπει να ισχύει και εντός των θεσμικών οργάνων. Συχνά βλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά απέναντι στους ε, καταγγέλλοντες. Οι άνθρωποι οι οποίοι ρισκάρουν τη ζωή τους για το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να έχουν τη στήριξή μας και εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Ε, έχετε μία μπλε κάρτα. Την έχετε, κύριε Γιάβορο. Κύριε Τζεκόφσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ασκήσατε κάποια κριτική για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς προστατεύουμε τους ανθρώπους αυτούς. Τι πιστεύετε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύετε ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αλλάξει τη, τη νοοτροπία και τη στάση, ε, μας ε, για να μην εξωστρακίζονται τα άτομα αυτά πλέον. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει τι άποψη έχει. Από το παρελθόν βλέπουμε πως ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια πολιτική απόφαση για το τι γίνεται για την προστασία των καταγγελόντων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει και να είναι υπόδειγμα και για τα θεσμικά όργανα και πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια νέα οδηγία η οποία θα εγγυάται μια ελάχιστη προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη. Για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας, ε, ο κ. Τζέιμς. Η κυρία Οι καταγγελίες, ναι, είναι δύσκολο θέμα δεδομένης της ερμηνείας και της διακριτικής ευχέρειας που υπάρχει. Είναι αποκάλυψη ή είναι εκδίκηση. Όσο πιο μυστικοπαθές ε, είναι ένα κράτος, ε, τόσο πιο επίμαχο γίνεται το ζήτημα. Είναι δύσκολο βεβαίως το ζήτημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε ήδη μια νομική κουλτούρα που διευκολύνει τις καταγγελίες, αλλά για πολλά άλλα κράτη-μέλη είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρείται ότι πηγαίνει κόντρα στον κρατικό μηχανισμό. Δεν πιστεύω πως η Κομισιόν έχει εδώ πέρα κάποιο ρόλο και άκουσα κάποιες εκκλήσεις για κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υιοθετηθεί κάτι τέτοιο και το έχουμε δει και σε άλλους τομείς. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους στην αίθουσα, όσο λίγοι και αν είναι, πως ε, οι πολίτες ε, των προεκομμουνιστικών χωρών θυμούνται ακόμα να τους χτυπάει κάποιος άγνωστος ε, την πόρτα με στη νύχτα και αυτό κατόπιν καταγγελίας. Έχουμε λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να μπλέκουμε με άσχετες υποθέσεις και δεν νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανένα ρόλο εδώ πέρα. Ευχαριστώ, Μπόνι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτοί που μας προειδοποιούσαν για πιθανούς κινδύνους πάντα ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για την κοινωνία, ειδικά τώρα που έχουμε πολλές διόδους πληροφορίας. Αν μας ειδοποιούν οι καταγγέλλοντες για διαφθορά, για παρανομίες έχουν και μια παρόμοια λειτουργία θα έλεγα με τους δημοσιογράφους που μας προειδοποιούν μέσω των ΜΜΕ. Και έτσι ο ρόλος τους είναι θετικός σε μια δημοκρατική κοινωνία. Όπως αναφέρθηκε στην έκθεση για την διαφθορά, υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα, καθώς υπάρχει μια προθυμία να κινηθεί κανείς κατά του οργανισμού του και για λόγους ε, αντεκδίκησης. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ακολουθούν την συνείδησή τους αλλά εκτός νομικού πλαισίου αναγκάζονται να παραβιάσουν τον νόμο για να ακολουθήσουν την συνείδησή τους όπως είπαμε. Και έτσι συνεισφέρουν στους δημοκρατικούς μηχανισμούς και αποκαλύπτουν εγκληματικές δραστηριότητες παραδείγματος χάρη την διαφθορά. Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγήσει στην καταστροφή του κράτους και της ε, λειτουργίας του. Σε δημοκρατικές κοινωνίες, παραδείγματος χάρη, οι δημοσιογράφοι έχουν δικαιώματα και προστατεύονται. Γι' αυτό πιστεύω πως πρέπει να αναπτύξουμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό και να προωθήσουμε την ενημέρωση για το θέμα, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βρεθεί ένα πλαίσιο για να προστατευτούν τα δικαιώματά τους ε, ως άτομα, ως επαγγελματίες. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει ήδη. Οπότε αυτό είναι καθήκον για όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σλέιν. Σλέιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι καταγγέλλοντες παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του οργανωμένου εγκλήματος, στη διαφθορά ε, εγκλήματα τα οποία γίνονται χαλαρά και άνετα και κινούνται και αψηφούν τα σύνορα. Είναι ευρωπαϊκά φαινόμενα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν ευρωπαϊκές λύσεις. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίσει τα ελάχιστα πρότυπα προστασία των καταγγελόντων για να μπορούν με κάθε ασφάλεια να αποκαλύπτουν τι πληροφορίε. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε δίθεν αυτά τα φαινόμενα, αλλά δεν προστατεύουμε αυτού που μιλάνε. Μόνο 8 ε, ευρωπαϊκά κράτη έχουν νομοθεσία για το θέμα. Το 2013 το Κοινοβούλιο, ε, στα πλαίσια της έκθεσης ΚΡΙΜ, ζήτησε με μεγάλη πλειοψηφία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2000, μέσα στο 2013 να περάσει μια νομοθετική πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος αποτελεσματικού και σφαιρικού για την προστασία των καταγγελόντων. Πέρασαν τρία χρόνια και δεν έχουμε δει ούτε μία λέξη την πρόταση αυτή. Ζητάω να μου πει η Κομισιόν γιατί αυτή η καθυστέρηση, γιατί αυτή η αντίσταση. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι από τον Ιανουάριο του 2014 τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κατέστησαν υποχρεωτική την εισαγωγή εσωτερικών κανόνων σε ό,τι αφορά τι καταγγελίες παρατυπιών. Εδώ ε, συμπεριλαμβάνουμε και την προστασία των πληροφοριοδοτών. Εκτός από το ελεγκτικό συνέδριο, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκαναν ελάχιστα για την προστασία των καταγγελόντων. Έτσι χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία για να δείξουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπέρ τη διαφάνειας και προστατεύουν αυτού που καταγγέλνουν τις παρατυπίες, τις αθέμητε και εγκληματικέ συμπεριφορέ. Ο κ. Χρυσόγονο. Η Ένωση οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των ανθρώπων που βοηθούν με τι πληροφορίε του να αποκαλυφθούν σκάνδαλα διαφθοράς σύμφωνα με έρευνα του 2013 της διεθνούς διαφάνειας οι περισσότερες χώρες της ένωσης αδυνατούν να προσφέρουν επαρκή νομική προστασία από αντίπεινα στον χώρο εργασίας ενώ η ανησυχία για ποινικέ διώξεις αποτελεί έναν ακόμα ανασταλτικό παράγοντα για τους πληροφοριοδότες. όπως παραδέχθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής ο κ. Γιούνκερ, το σεπτέμβριο του 2015 ενώπιον του ευρωκοινοβουλίου πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο ζήτημα αυτό. Α αναλογιστούμε όλοι τις διαστάσεις του σκανδάλου luxleaks ή του σκανδάλου volkswagen και θα αντιληφθούμε πόσο θα βοηθούσε αν υπήρχε εναρμονισμένη νομοθεσία ώστε οι πληροφοριοδότες να μην φοβούνται να καταγγείλουν όσα γνωρίζουν. η διαφθορά κινείται στο σκοτάδι. μόνο αν δώσουμε κίνητρα στους πολίτες να βγουν στο φως και να την καταγγείλουν θα μπορέσουμε να την καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά. ευχαριστώ. parola, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το ΕΛΚ είναι πεπισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αξίες όπως είναι η διαφάνεια, η ακαιρεότητα και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σε όλους εκείνους οι οποίοι αποφασίζουν να καταγγείλουν παραβιάσεις τέτοιων αξιών. Όσοι λοιπόν χτυπούν το κουδούνι του συναγερμού βοηθούν να διασφαλίσουμε ότι δεν γίνεται κατάχρηση από αυτούς που δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός αυτός υπάρχει, προστατεύεται και αυτό έχει να κάνει και με τον κύριο Χασάν τον ίδιο. Παρά τις προσωπικές μου επιφυλάξεις για την προσωπικότητα του κύριου Ασάνς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το τι έκανε, γιατί αυτό που έκανε μας επέτρεψε να καταλάβουμε πόσο περίπλοκα είναι κάποια διεθνή ζητήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τάση να κρύβουν τα πράγματα κάτω από το χαλί. Αλλά άλλοι, σαν τον κύριο Ασάνς, δεν το κάνουν. Δεν βολεύονται έτσι. Είναι λοιπόν ε, κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και ότι οι άνθρωποι αυτοί συχνά γίνονται θύματα στο τέλος. Εμείς λοιπόν οι ευρωβουλευτές, οι εκπρόσωποι του κόσμου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο. Πιστεύω λοιπόν ότι η φυλάκιση του Ζουλιάν Σανς πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να προσφέρουμε διεθνή νομική προστασία. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασφαλίσει επαρκή προστασία στον Ασάνζο και στους άλλους καταγγέλλοντες, αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό μήνυμα που στέλνουμε σε όσους είναι διατεθειμένοι να κάνουν τέτοιες καταγγελίες. Ο κύριος Φλάναγκαν. Όπως τόσοι οι άλλοι και τόσα άλλα θέματα, έτσι και εδώ καθόμαστε και συζητάμε για ένα θέμα όπου η πραγματικότητα είναι κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που συζητάμε εδώ. Πριν από 8 χρόνια ο Σούκαμαν παρετήθηκε από τη δουλειά του που ήταν manager στην Unicred τη Ιρλανδία. Είπε ότι το έκανα αυτό για να μην βρεθώ εγώ στη θέση του εγκληματία. Επρόκειτο για θέματα οικονομικά της τράπεζας και αυτά που είπε ότι έβλεπε κάθε μέρα ήταν ότι η τράπεζα δεν είχε τα χρήματα τα οποία έλεγε ότι είχε. Και δεν μιλάμε τώρα για δεκαδικά, αλλά μιλάμε για 40 φορές παραπάνω όσον αφορά την νομοθεσία. Τώρα τα είπε. Τα είπε στους ρυθμιστές της τράπεζας. Η τράπεζα του είπε πάψε μη λες τίποτα. Ε, προσπάθησε να προχωρήσει για να υπάρξει έρευνα, αλλά του είπαν ότι δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει ότι θα έχει ασυλία ή την ακαιρεότητά του. Δεν του ζήτησαν καν τελικά όταν έγινε έρευνα για την τράπεζα να πάει ως μάρτυρας. Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για αυτά όταν έχουμε καταγγέλλοντες και δεν τους προστατεύουμε σημαίνει ότι κάτι έχουμε να κρύψουμε. Πρόεδρε, όταν μιλούν εδώ κάποιοι μπορούν αυτοί που κάθονται κοντά τους να μην μιλάνε στο τηλέφωνο γιατί τους ενοχλούν και γιατί δεν τους παρακολουθούν. Mm. Ευχαριστώ. Θεωρώ τη συζήτηση αυτή για τους καταγγέλλοντες σαν ένα μέτρο κατά της διαφθοράς και μάλιστα ένα στοιχείο κλειδί κατά της διαφθοράς. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στις χώρες μέλη. Ο Ευρωπαίος πολίτης θεωρεί τη διαφθορά σαν ε, ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που τον απασχολούν. Στις περισσότερες χώρες ε, μέλη δεν υπάρχει ρύθμιση επαρκής για την προστασία των καταγγελόντων μόνο σε κάποιους κώδικες εργασίας ε, χωρών μελών κάτι αναφέρεται. Οπότε κύριε Επίτροπε θα πρέπει να σκεφτείτε πώς μπορεί να υπάρξει μια γενική ρύθμιση που θα καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας για τους καταγγέλλοντες. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, οδηγιών όπου κάτι αναφέρεται για τα άτομα αυτά. Όμως μια γενική ρύθμιση αξίζει τον κόπο αν δίνει μια ελάχιστη προστασία σε περίπτωση εγκλημάτων, σοβαρών εγκλημάτων και όχι μόνο τα πρόκειται για ηθικά ζητήματα. Όπως έχει σήμερα η νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Είναι και αυτό μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Πριν από μερικά χρόνια ήμουνα υπεύθυνο αυτή της προβληματικής στην Τσεχία όταν ήμουν υπουργό εκεί. Δεν υπήρχε όμως παρκή πολιτική βούληση για να υιοθετηθεί τέτοια νομοθεσία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα ήταν καλό τέτοια νομοθεσία να υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προστατευτούν αυτοί που δεν φοβούνται να καταγγείλουν παρατυπίες. Ευχαριστώ. Κάτσε τη τώρα. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσοι λίγοι τολμούν να καταγγείλουν παρανομίες δεν την χάνουν επαρκούς νομικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά παρότι οι καταγγελίες έχουν καταδείξει τη χρησιμότητά τους αφού τα διάφορα τραπεζικά σκάνδαλα τα σκάνδαλα τύπου volkswagen το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η φοροδιαφυγή και η αποφυγή είναι στην ημερήσια διάταξη. το σκάνδαλο των luxleaks οι λίστες borgens και lagarde που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως από τις αρμόδιες αρχές ιδίως στην ελλάδα έδειξαν ότι φυσικά πρόσωπα αλλά και πολυεθνικές συστηματικά φοροδιαφεύγουν και φοροαποφεύγουν. η θέσπιση λοιπόν της προστασίας των καταγγελόντων παρανομίες είναι βέβαιο ότι θα αναδείξει και άλλες περιπτώσεις παραβίασης της φορολογικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας των κρατών της ευρωπαϊκής ένωσης εν γέννη είναι λοιπόν προ όφελο των ευρωπαίων πολιτών να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο προστασία αυτών των ανθρώπων. δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε πρόεδρε τι πρόσφατε διώξει κατά δημοσιογράφων στο λουξεμβούργο που αποκάλυψαν το σκάνδαλο των luxleaks. ευχαριστώ. Ε. Και τώρα, ο κύριος Ανδρουκάητης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα καταληκτικά λόγια. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, την άκουσα μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ θερμά τους συμμετέχοντες στη συζήτηση αυτή. Θα ενημερώσω τους συναδέλφους μου τον αρμόδιο επίτροπο που είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Και θα του πω ότι του είπατε. Συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες. Το θέμα είναι πώς. Δηλαδή, τι είναι καλύτερο να κάνουμε και τι είναι ρεαλιστικό να κάνουμε. Το θέμα είναι φυσικά πολύ περίπλακο. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχουν δυνατότητες να φτιάξουμε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο για να τους προστατεύσουμε. Ο Αρμόδιος Επίτροπος μου είπε να σας στείλω το εξής μήνυμα. Επιθυμεί να συνεχίσει τις συζητήσεις μαζί σας, να εμβαθύνουμε στον προβληματισμό και σας ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Έκλεισε η συζήτηση.